έχει ζητήσει διόρθωση σε κείμενο του Κοινοβουλίου βάσει του άρθρου 231 παράγραφος 4 του κανονισμού αυτή η διόρθωση θεωρείται εγκεκριμένη εκτός και ε, σε 24 ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας πολιτική ομάδα ή ομάδα αριθμός βουλευτών ίσως με το ελέγχιστο όριο δεν εκφράσουν αντίρρηση ε, το διορθωτικό στο κείμενο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Ολομέλειας και ο τίτλος του θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της τρέχουσας Ολομέλειας. Ήθελα επιπλέον να ενημερώσω την Ολομέλεια ότι μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου